Uh, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε το σκέλος ε, της ΕΚΟΝ. Ένα σημείο έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση, παρουσίαση, έκθεση τέλο πάντων, την οδηγία για τα MPL. Μη εξυπηρετούμενα δάνει. Κυρία Ντελάγκη, θέλετε να ξεκινήσετε, Εστέρ. Uh, uh, Μετά από την υπερδιέγερση έχουμε χαλαρώσει λίγο, λοιπόν πάρα πολύ σύντομα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καταφέραμε να συμφωνήσουμε, όπως είχαμε υποσχεθεί, ε, σε μια κοινή θέση πριν τις εκλογές για ένα τεχνικό και λεπτό ε, θέμα αφού πρώτα συμφωνήσαμε και σε ό,τι αφορά το εποπτικό backstop θα ψηφιστεί αργότερα αυτήν την εβδομάδα στην Ολομέλεια. Η δική μας δουλειά ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή ΕΚΟΝ, ως ενισηγητές, ήταν να έχουμε μια φιλόδοξη οδηγία για την ευθερογενή αγορά NPL. Υπήρχαν διάφορα συμφέροντα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κράτη-μέλη, τους καταναλωτές, ε, τους συμμετέχοντες στην αγορά. Θέλαμε την αρχή λοιπόν να τα καταφέρουμε σωστά. Είχαμε ε, κάποιες βάσεις και κάποιες αρχές εργασίας, διασυνοριακές δραστηριότητες περισσότερο για χώρες που έχουν υψηλά αποθέματα μη δανείων, ε, για τις ΜΜΕ, για τους καταναλωτές, ειδικέ ασφαλιστικές κλίσεις αυτό το είχαμε συστήσει και στους σκιώδες εισηγητές. Επίσης θέλαμε ε, να μην παραφορτώσουμε το νομικό σύστημα των κρατών μελών. Θέλαμε έξτρα ασφαλιστικέ δικλείδε για το ξέπημα χρήματο και πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο ήδη ε, σε αυτή τη θητεία. Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Και τις αρχές αυτές ε, τις σεβαστήκαμε για κάποια βασικά ζητήματα να πω. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, το σχέδιο έκθεση έχει μια πολύ στοχευμένη προσέγγιση. Περιορίζει το πεδίο εφαρμογή μόνο ε, σε μη εξυπηρετούμενε συμφωνίε μεταξύ διαχειριστών και αγοραστών πιστώσεων υπήρξε ένα πιθανό πρόβλημα σε ό,τι αφορά ε, τη δυνατότητα να συνεχίζουν οι διαχειριστές πιστώσεων τις αστηρότητές ε, τους σε κάποιες προϋποθέσεις το λύσαμε υπό κάποιες συνθήκες, ε, λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, η προστασία των καταναλωτών, παραλαμβάνω το ένα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα διαβατηρίου για τους αγοραστές ε, παραμένουν. Αυτό το άρθρο 11, ένα άλλο σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής αλλαγή των όρων ε, του δανείου. Αυτό το είχαμε συζητήσει με τους κοιόδης. Επίσης, ότι αφορά τις απαιτήσει περιπληροφόρηση και για τους αγοραστές και για τους δανειολήπτους. Στο άρθρο 13 τις έχουμε επεκτείνει και για τα κράτη-μέλη, γιατί για κάποιους από εσάς ήταν πολύ σημαντικό, ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να υπερβούν ε, και να έχουν πιο αναλυτικούς όρους και πιο διεξοδικούς. Για το άρθρο 5 δεν θέλουμε να πέσει τον κάλτο να αχρήστων. Θέλαμε όμως μια γρήγορη συμφωνία. Γι' αυτό έχουμε το δεύτερο τμήμα ε, που θα το δούμε αργότερα. Χωρίσαμε στα δύο δηλαδή. Ευχαριστώ και το συνεισηγητή και όλο το προσωπικό για την πολύ καλή συνεργασία. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τη συνεισηγητρία. Ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα γιατί είναι πολύπλοκο το κείμενο και έπρεπε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Δεν ήταν και εύκολο αυτό, αλλά νομίζω το καταφέραμε. Έχουμε λοιπόν τώρα το δεύτερο δομικό, ας πούμε το δεύτερο ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής για τη μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με πρώτο ακρογωνιαίο λίθο το εποπτικό backstop. Να πω εγώ που χρειάζονταν βελτιώσεις σε σχέση με το κείμενο ε, πολύ χαμηλό επίπεδο αστικά κοινών απαιτήσεων. Και τα κράτη-μέλη αστικά ήταν αυτά τα οποία ε, θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Βέβαια είχαμε έναν κανονιστικό υπερθεματισμό. Δεν ήταν και το ιδεώδες. Εμείς θέλαμε πιο απαιτητικούς όρους και απαιτήσει για διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων. Ζητήσαμε λοιπόν πιο αυστηρές οι απαιτήσει. Ιδίω για τη ρευστότητα, για του ίδιου πόρους, τη διακυβέρνηση, ε, την προστασία των δανειοληπτών, προστασία δεδομένων και άλλα μέτρα για τη διαχείριση αναφορά κινδύνων, επίσης ξέπλυμα χρήματος και αντιμετώπιση τρομοκρατίας. Εμεί δηλαδή ουσιαστικά ακολουθήσαμε τον τρίτο δρόμο. Αφενό είχαμε τις ελάχιστες κοινέ απαιτήσει και από την άλλη είχαμε ε, μια προσέγγιση που θα άφηνε στα στις εθνικές αρχές ε, τη διακριτική ευχαίρεια και εμεί είμαστε κάπου στη μέση. Η δεύτερη δυναμία, κατά την άποψή μου, στην πρόταση της Κομισιόν ήταν ένας κίνδυνος που διέβλεψα. Να έχουμε ένα, ένα μοντέλο αναδυναμητικό που οι τράπεζες θα ελέγχουν τη φερεγγιότητα ε, και θα περνάνε τον κίνδυνο σε άλλο φορέα. Θέλαμε λοιπόν και αποφασίσαμε να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μόνο, γιατί η αρχή πρόταση είχε ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Και αυτό ευθυγραμμίζεται και με το έργο του Συμβουλίου. Και ένα τρίτο στοιχείο, σε σχέση με τη δεύτερη πάντα δυναμία, για να έχουμε αποτελεσματική προστασία των δανειοληπτών και να προστατεύσουμε και την δευτερογενή αγορά. Οι αγοραστές πιστώσεων υποχρεούνται να ε, προσφεύγουν σε πιστοτικούς ε, φορείς διαπιστευμένους, είτε πιστοτικά εντρήματα είτε εχειριστές πιστώσεων. Έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε και τους καταναλωτές αλλά όλους τους δανειολήπτες επίσης και τις ΜΜΕ. Τέλος, επειδή η εποπτεία και επιβολή κυρώσεων με εξοδεδομένων φορέων όπως αγοραστών ε, πιστώσεων θα ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό, άρα δεν θα ήταν και αποτελεσματικό, επιβάλλουμε στους ε, διαχειριστές πιστώσεων όλες τις απαιτήσει. Ε, με αυτή την τροπολογία νομίζω διευκολύνεται το συνολικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξήγησα το λόγο για τον οποίο Την εξοδικαστική επιβολή για τα θέματα των ε, εγγύσεων Το αφήσαμε εκτός γιατί θέλαμε να προχωρήσουμε με το φάκελο αυτό. Οπότε διαγράφει αυτό το σκέλος της πρότασης της Κομισιόν για το ICE. Θέλαμε λοιπόν να έχουμε μία ε, δευτερογενή αγορά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελεσματική, αλλά ταυτόχρονα χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ύψη στο επίπεδο προστασία των καταναλωτών και δανειοληπτών εν γέννη. Άρα, νομίζω με την έκθεση αυτή έχουμε βρει τη χρυσή τομή, ε, τη σωστή ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των στοιχείων και οι τρει συνιστώσει και τα τρία σκέλη για μένα είναι ουσιώδη για μια μελλοντική συμφωνία με το Συμβούλιο που ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα. Αν βέβαια και εμείς προχωρήσουμε γρήγορα, ε, γκρίνοντας αυτό το κείμενο. Φυσικά θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τις τροπολογίες και θα λάβουμε υπόψη τις παρεμβάσεις και τις ε, γραπτές παρατηρήσεις όλων των σκιωδών. Και περνάω τώρα στους σκιώδεις. Ο Μπέρντ Λούκε είναι ο πρώτος. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές ε, για την ε, έκθεση αυτή. Έχουμε χείρας και χαίρομαι ε, που άκουσα και από το στόμα του Ρομπέρτο. Ότι έχετε στόχο να εξετάσετε πολύ προσεκτικά και να μελετήσετε τις τροπολογίες και ε, όταν είδα το χρονοδιάγραμμα είχα τις αμφιβολίες μου για το κατά πόσο αυτό θα ήταν εφικτό ε, σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Χαίρομαι και ελπίζω τα λόγια να γίνουν και έργα, ώστε να μπορέσουμε πράγματι να ολοκληρώσουμε εγκαίρως. Σε ό,τι αφορά του συνεισηγητέ, ε, σε ό,τι αφορά τα εξοδικαστικά, είπατε ότι θα τα αφήσετε εκτός. Ε, είναι ένα επίμαχο ε, σημείο, έγινε επίμαχο, οπότε μάλλον είναι καλό που το αφήσαμε κατά μέρος προς το παρόν ε, το θέμα αυτό για τις εγγύσεις. Τώρα, ένα θέμα το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι τα δικαιώματα και προστασία των καταναλωτών και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό τα δικαιώματα των καταναλωτών να γίνονται σεβαστά και στο μέλλον. Και να ε, μην επερέχουν, ε, υπερτερούν τα δικαιώματα των ε, τραπεζών, τα αρχικά δικαιώματα. Αν δηλαδή σε ό,τι αφορά την παραχώρηση της πίστοσης αυτής σε έναν servicer, σε έναν διαχειριστή. Να μην υπάρχει δηλαδή μικρότερο recovery rate για τον Credit Service Provider. Ähm, äh, Γιατί αυτό ε, τελικά θα δημιουργήσει ε, υψηλότερους ε, συντελεστές και για τους υπόλοιπους να δανειολήπτες. Ε, οπότε πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα δικαιώματα των καταναλωτών σε αυτήν την περίπτωση και πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά ε, να ε, ορίσουμε τις διτάξεις της οδηγίας ώστε να ενισχύονται ακόμη περισσότερο αυτά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα καταθέσω σχετικά και τροπολογίες και θα τα πω και στους άλλους κοιόδες της συνεδρίας. Νομίζω όμως ότι η πρόταση είναι καλή, είναι μια καλή βάση συζήτηση και προσβλέπω και στην καλή συνεργασία με τους συναδέλφους. Uh, uh, Ευχαριστούμε για την ALDE, ο Ραμόν Τρεμόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακόμη και αν δεν μας αρέσει η οδηγία αυτή, δημιουργεί διχασμό, αλλά θα πρέπει το, ισχυρό, το, μήνυμα του Κοινοβουλίου να είναι ισχυρό και να ε, οδηγήσει και σε ένα σαφέ συμπέρασμα ε, τη εργασία του Συμβουλίου. Γι' αυτό θα πρέπει να να επιζητήσουμε την ε, ανάκτηση των εγγύησεων. Η στάση της ομάδας έχει να κάνει με το πώς οι δευτερογενείς αγορές μπορούν να αλλοιώσουν τη φύση των NPL και να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών μέσων, όπως είπε προηγουμένω και ο Μπεν ε, και αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που προσπιστήκαμε και στο προηγούμενο θέμα, γι' αυτό που βάλαμε σχετικά τροπολογίες που ελπίζουμε θα το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. για τη βαθμία μείωση των MPL. Είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκέ αρχέ που παρακολουθούν, που πτεύουν τι ε, αγορέ αυτέ, να μπορούν να επιβάλλουν αυτό το νομικό πλαίσιο, να το εφαρμόσουν, για να μην υπάρξουν ατασταλίε και εκτροχιασμοί λόγω ε, διαφορετική μεταφορά τη εθνική νομοθεσία. Γι' αυτό θέλουμε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η EBA, να έχει λόγο εδώ. Διότι οι αρχές των κρατών που θα είναι αρμόδιες θα παρακολουθούν τους ε, πιστωτές και πολίτες, αλλά γιατί να μην δώσουμε και στην EBA ε, τη δυνατότητα να παρακολουθεί αυτούς που παρακολουθούν. Η EBA λοιπόν αναλάβει εδώ ένα σημαντικό ρόλο. Διότι όταν ε, χρησιμοποιείται μια νομοθεσία από το Κοινοβούλιο, όταν προτείνεται μια νομοθεσία από το Κοινοβούλιο, πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί και από τα κάτι μέλη. Κοιτάμε λοιπόν τι γίνεται στι ευρωπαϊκέ αγορέ για να εφαρμόσουμε τι φέλτιστε πρακτικέ. Όχι να έχουμε ε, τι ε, αποκλίνουσε συμπεριφορέ που βλέπουμε στα διάφορα κάτι μέλη. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε στι ευρωπαϊκέ αρχέ για να έχουμε ίσους κανόνε παιχνιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τους πράσινους ο κύριος Ουρτασούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τους πράσινους ένα σχόλιο μόνο για τη μεθοδολογία. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Διότι μόλις πριν τη συζήτηση λάβαμε την τελευταία εκδοχή της πρότασης. Δεν βοηθάει πολύ ε, θέλουμε να υπάρχει μια μεγάλη συμμαχία και στήριξη για την έκκληση γενικώ, αλλά αν θέλετε από τη δική μα την ομάδα στήριξη, θα πρέπει να μα δώσετε λίγο χρόνο για να το μελετήσουμε το θέμα. Είναι και θέμα του ρυθμού τη δουλειά μα τι επόμενε μέρε. Ω προ το περιεχόμενο, να πω ότι σε αντίθεση με του εξωτερικού μεταρρυθμιστέ, Χαιρόμαστε που ασχολούμαστε μόνο με τις διευθετήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αυτό είναι το σημαντικό, αλλά και οι δανειστικές υπηρεσίες θα πρέπει να συνεχιστούν ε, βάσει της οδηγίας αυτής, αναπερίπτωση, και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εφόσον αυτά μπορούν τελικά να αποπληρώνονται. Ίσως χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις από την πλευρά σας για το σημείο αυτό. Επιπλέον, θέλαμε πιο συγκεκριμένε υποχρεώσεις για τους προστατές που ασκούν λογική λογικά, ε, που επιβάλλουν λογικούς κανόνες σε αυτούς τους μη εξυπηρετούντες ε, για την αποφυγή της πώληση των εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτα μέρη. Στην παρουσίασή σας επίση ακούσαμε ότι θέλετε αυστηρότερες ε, προποθέσει για τις επιστατικές υπηρεσίες όπως προτείνει και η πρόταση τη Κεντρική Τράπεζα. Το στηρίζουμε αυτό. Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέλλον το στηρίζουμε αυτό. Αλλά ένα μεγάλο μέρο των επιστοτικών υπηρεσιών ε, δεν καλύπτουν αυτού του κανόνε, όπω τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα επενδυτικά ταμεία. Αυτό είναι επίση ένα θέμα για μα. Γιατί περιορίσατε το πεδίο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα καλύπτουν την οδηγία, διότι και αυτό μα ανησυχεί. Επιπλέον, απαιτήσει ίσω είναι αυστηρέ, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν με λεπτομερεί υποχρεώσει για την ε, ε, δέουσα και ταχεία ε, εκπρέτηση των πιστωτών με ένα ενιαίο νομοθέτημα που να αφήνει όλους τους όσους λειτουργούν στην αγορά αυτή στην, στον ύκτο των απαιτήσεων της EBA. Θα πρέπει επίσης οι υπηρεσίες να προσφέρονται ανάλογα με το τι κανόνες προσ... προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία του κάτους μέλους υποδοχή, ανάλογα με το άρθρο 139 και στο 135 ε, όπου εξελίσσεται η αρμοδιότητα των, αρχών, των αρμόδιων αρχών του κράτους υποδοχής να, προ... να απαγορεύσουν υπηρεσίες και την προσφορά τους σε αυτό το κάτο μέλος, το οικείο κράτος μέλος, μέχρι να ληφθεί η απόφαση για την προσφορά υπηρεσιών τη συγκεκριμένη και αυτό είναι κάτι που μας αρέσει. Και εδώ ε, πρέπει να δούμε τη δευτερογενή αγορά μέχρι να δούμε κατά πόσον μπορούν να παρέμβουν οι τράπεζες στην πώληση του χαρτοφυλακίου σε ένα τρίτος μέρος. Thank you. Um, e. Κύριε θα ήθελα να... Ε, θα ήθελα ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για την ε, δουλειά που μας παρουσίασαν. Άκουσα με ενδιαφέρον ότι θα εξετάσετε και θα αξιοποιήσετε τις τροπολογίες που θα κατατεθούν, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη γιατί το χρονοδιάγραμμα που μας παρουσιάσατε μας δίνει ελάχιστες μέρες να καταθέσουμε προτάσεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις. Θα επιδιώξουμε τη βελτίωση αυτού που έχουν συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με την ομάδα των σοσιαλιστών και μένει και εσείς να αποδείξετε ότι δεν έχετε μια προκατασκευασμένη συμφωνία ανελαστική όσον αφορά την αποδοχή άλλων προτάσεων. Επειδή η ώρα είναι προχωρημένη, θα είμαι σύντομος. Οι τροπολογίες που θα καταθέσω εξ ονόματος της Ευρωομάδας της Αριστεράς θα επιδιώξουν να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών μέσα από ένα αριθμιστικό πλαίσιο υπερασπίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα γιατί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ τελευταία φορά που λογαριάστηκαν συνολικά, αλλά χωρίς να υπερβαίνουμε την αρχή της αναλογικότητας σε βάρος της προστασίας του καλώς εννοούμενου δημοσίου συμφέροντος και των καταναλωτών. Άρα η πρώτη επιδίωξή μας μέσα από τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε είναι να ενισχύσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει τους καταναλωτές απέναντι σε καταχρήσεις δύναμης και εξουσίας. Και ένα δεύτερο, είναι ότι για αυτή τη δευτερογενή αγορά που δημιουργείται έχει ιδιαίτερη σημασία οι εξωτερικές πιστοτικές υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το outsourcing, θα πρέπει να υπόκειται σε έναν διαφανή δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία για λόγους υπεράσπισης όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος. Αυτό που θα φανεί στην πορεία είναι, κύριε Πρόεδρε, ε, εάν θα δεχθείτε κάποιες από τις προτάσεις που θα καταθέσουμε εμείς ή ε, άλλες πολιτικές ομάδες μέσα από τις τροπολογίες μας ή αν έχετε μία ανελαστική συμφωνία την οποία μας παρουσιάζεται εδώ με σκοπό να την επιβάλλετε κατά πλειοψηφία. Uh, Σας ευχαριστούμε. Ε, όπως και οι προηγούμενοι συναδελφοί μου, ανησυχώ κάπως το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο δεν αφήνει να το συζητήσουμε. Δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε τη διερμηνία διότι το προβλεπόμενο τέλος είναι στις 9. Δυστυχώς θα πρέπει να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα